Τι τώρα στα πολεμικά συνεχίζω πρώτα να σας ανακοινώσω τώρα τα αποτελέσματα των εκλογών για τους αντιπροέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, ψήφισαν 701 βουλευτές στι εκλογές και είχαμε 17 ψήφους άκυρες. Άρα 684 ήταν οι έγκυρες ψήφοι, η δε απόλυτη πλειοψηφία είναι 343 ψήφοι. Τώρα, έκαστος των υποψηφίων έλαβαν ε, έλαβε τις εξής. Αντζελίλη, 277 ψήφους. Ιζαμπέλ Ντιρόν, 268. Καμίνσκι, 194. Κοχ Μέρλιν, 148. Κράτσα Τσαγκαροπούλου. 355. Σταύρος Λαμπρινίδης. 348 ψήφους. Μακμίλαν Σκότ. 237 ψήφους. Μιγγέλ Άγγελ Μαρτίνεθ Μαρτίνεθ. 330. Πιτέλα. 360 ψήφους. Ροτ Μπέρεντ. 299. Λίμπορ Ρότζεκ. 284. Παλ Σμιτ. 266. Βιντάλ, Κουάδρος 332 303 ο Wallace ο κύριος Βίλαντ 267 οι εξή υποψήφοι έλαβαν την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων Πιτέλα Κράτσα Τσαγκαροπούλου και Σταύρο Λαμπρινίδης θα πρέπει να συγχαρώ αυτούς τους υποψηφίους Jedenaście miejsc jedenaście miejsc w ramach wyboru wiceprzewodniczących pozostaje do obsadzenia. Należy zatem przystąpić do drugiej tury. Έχουμε 11 θέσει των που θα πρέπει να καλυφθούν. Επομένω, θα πρέπει να γίνει τώρα ο δεύτερο γύρο ε, ε, τη ψηφοφορία. Εάν επομένω δεν έχουμε κάποια ένσταση, κάποια παρατήρηση, τότε θα ε, κρατήσουμε το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου. Ε, οι υποψήφοι που εξελέγησαν ε, θα συνεχίσουν και έχουμε μια διακοπή 10 λεπτών. Διακόπτουμε 10 λεπτά για να πάρετε τα ψηφοδέλτια. Διακοπή 10 λεπτών. Παρακαλώ μην φεύγετε από την αίθουσα. It was no probably translation. Please stay here in the... Επαναλαμβάνει στα αγγλικά. Μάλλον δεν μεταφράστηκε. Παρακαλώ μείνετε στην αίθουσα. koleżanki i koledzy wznawiam posiedzenie wznawiam posiedzenie powtarzam And... Αγαπητοί συνάδελφοι, σας παρακαλώ ακούστε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα σας πω. Θα απαιτηθεί τρίτος γύρος ψηφοφορίας. Οπότε σας παρακαλώ μην φύγετε από την αίθουσα γιατί στις 7.30 θα ακολουθήσει τρίτος γύρος ψηφοφορίας. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ζητήσω από τους καταμετρητές των ψήφων να καταλάβουν τις θέσεις τους και αυτοί θα ψηφίσουν τελευταίοι σας έχουν το δοθεί ψηφοδέλτια. Σας παρακαλώ λοιπόν χρησιμοποιήστε μόνο αυτά τα ψηφοδέλτια. Βάζετε ένα σταυρό δίπλα στο όνομα του ατόμου που επιθυμείτε να ψηφίσετε. 11 θέσεις πρέπει ακόμα να πληρωθούν. Επειδή λοιπόν 11 είναι τα άτομα, 11 σταυρούς μπορούτε, μπορείτε να βάλετε. Σας επαναλαμβάνω λοιπόν και στα αγγλικά μόνο 11 άτομα μπορείτε να ψηφίσετε. Στην περίπτωση που θέλετε να κάνετε κάποια διόρθωση, παρακαλώ απευθυνθείτε στους κλητήρες να σας δώσουν καινούριο ψηφοδέλτιο και το παλιό θα καταστραφεί. Άρχεται η ψηφοφορία. Yes, 90, okay. Uh, well, it is 90. Okay, okay. Uh, Mr. Colleague Leichtfried, please take the floor. Παρακαλώ. Έχετε... Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ε, παρέμεινε η ερώτησή μου μετά από αυτές τις ε, λεπτομερείς εξηγήσεις που δώσατε. <laughs>